Αρχίζει η συνεδρίαση. Κατόπιν διαβουλεύσεων με τις πολιτικές ομάδες θα ήθελα να σας ενημερώσω για τις ακόλουθες αλλαγές στην ημερήσια διάταξη κατόπιν της ανακατανομής των ψηφοφοριών στις διαφορετικές διαδικασίες ψηφοφορίας οι τελικές ψηφοφορίες για το πακέτο κοινή αγροτικής πολιτικής εκθέσεις Γιάρ, Μιούλερ και Αντριέ μετακινούνται στη δεύτερη διαδικασία ψηφοφορίας της σημερινής ημέρας. Κατά συνέπεια, η τρίτη διαδικασία ψηφοφορίας που είχε προγραμματιστεί για σήμερα Παρασκευή 23 Οκτωβρίου από τις 18 στις 19 και 15 ακυρώνεται όπως και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στις 21 και 30. Οι επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τις ψηφοφορίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο τμήμα Σημαντικές πληροφορίες. Δεν βλέπω να υπάρχει κάποια αντίρρηση. Η αλλαγή εγκρίνεται θα ξεκινήσω με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της χθεσινής τρίτης ψηφοφορίας. Το αποτέλεσμα, τα αποτελέσματα της τρίτης ψηφοφορίας της 5ης 22 Οκτωβρίου έχουν ως εξή. Κοινή γεωργική πολιτική στήριξη των στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται από τα κράτη-μέλη και να χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΦΕ και από το εΓΤΑΦΑΛΦΑ. Τροπολογία 857 απορρίπτεται. Τροπολογία 1000 απορρίπτεται. Τροπολογία 796 εγκρίνεται. Τροπολογία 1001 απορρίπτεται. Τροπολογίες 1002 και 1183 απορρίπτονται. Τροπολογία 1003 απορρίπτεται. Τροπολογία 797 εγκρίνεται. Τροπολογία 858 εγκρίνεται. Τροπολογία 1004 απορρίπτεται. Τροπολογία 798 εγκρίνεται. Τροπολογία 799 <clears throat> απορρίπτεται. Τροπολογία 730 εγκρίνεται. Τροπολογία 800 πρώτο μέρος εγκρίνεται. Τροπολογία 800 δεύτερο μέρος απορρίπτεται. Τροπολογία 801 εγκρίνεται. Τροπολογία 859 απορρίπτεται τροπολογία 802 πρώτο μέρος εγκρίνεται τροπολογία 802 δεύτερο μέρος εγκρίνεται τροπολογία 803 εγκρίνεται τροπολογία 1144 πρώτο μέρος εγκρίνεται τροπολογία 1144 δεύτερο μέρος εγκρίνεται τροπολογία 860 απορρίπτεται κοινή γεωργική πολιτική, χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση. Τροπολογία της αρμόδιας επιτροπής ψηφοφορία κατά σύνολο εγκρίνεται. Τροπολογία 233 απορρίπτεται. Τροπολογία 207 απορρίπτεται. Τροπολογία 240 απορρίπτεται. Τροπολογία 76 εγκρίνεται. Τροπολογία 241 απορρίπτεται. Τροπολογία 77 εγκρίνεται. Τροπολογίες 79 και 242 εγκρίνονται. Τροπολογίες 243 και 245 απορρίπτονται. Τροπολογία 81 εγκρίνεται. Τροπολογίες 82 και 244 εγκρίνονται. Τροπολογία 246 απορρίπτεται. Τροπολογίες 84 και 247 εγκρίνονται. Τροπολογία 248 απορρίπτεται. Τροπολογία 249 απορρίπτεται. Τροπολογία 93 εγκρίνεται. Τροπολογία 250 απορρίπτεται. Τροπολογία 94 εγκρίνεται. Τροπολογία 251 απορρίπτεται. Τροπολογία 252 απορρίπτεται. Τροπολογία 257 απορρίπτεται. Τροπολογία 288 απορρίπτεται. Τροπολογία 289 απορρίπτεται. Τροπολογία 227 εγκρίνεται. Τροπολογίες 183, 211 CP1, 283 CP1 εγκρίνονται. Τροπολογία 290 απορρίπτεται. Τροπολογία 211 CP2 εγκρίνεται. Τροπολογία 283 CP2 απορρίπτεται. Τροπολογίες 184, 185, 186, 187, 188, και 211 CP3, 283 CP3 εγκρίνονται. Τροπολογία 292 απορρίπτεται. Τροπολογία 211 CP4 απορρίπτεται. Τροπολογία 291 εγκρίνεται. Τροπολογία 189. 211 CP5, 283 CP4 εγκρίνονται. Τροπολογία 283 CP5 απορρίπτεται. Τροπολογίες 190, 191, 211 CP6 εγκρίνονται. Τροπολογία 212 CP1 και 293 εγκρίνονται. Τροπολογία 212 CP2 και 294 εγκρίνονται. Τροπολογία 228 εγκρίνεται. Τροπολογίες 192 και 193 καταπίπτουν. Τροπολογία 213 απορρίπτεται. Τροπολογία 259 απορρίπτεται. Τροπολογία 258 απορρίπτεται. Τροπολογία 260 απορρίπτεται. Τροπολογία 298 απορρίπτεται. Τροπολογία 261 απορρίπτεται. Τροπολογία 262 απορρίπτεται. Τροπολογία 202 εγκρίνεται. Τροπολογία 230 εγκρίνεται. Τροπολογία 263 απορρίπτεται. Τροπολογία 264 απορρίπτεται. Τροπολογία 284 εγκρίνεται. Τροπολογία 208 καταπίπτει. Τροπολογία 1 καταπίπτει. Τροπολογία 231 απορρίπτεται. Τροπολογία 232 απορρίπτεται. Τροπολογία 13 εγκρίνεται. Τροπολογία 299 εγκρίνεται. Τροπολογία 209 και 285 εγκρίνονται. Τροπολογία 210 και 286 εγκρίνονται τροπολογία 30 καταπίπτει, τροπολογία 287 απορρίπτεται, τροπολογία 31 εγκρίνεται. Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά, ως τις 9 η ώρα. Έχουμε 7 λεπτά διακοπή. Σας ευχαριστώ. Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται. Θα προχωρήσουμε στη σημερινή πρώτη ψηφοφορία. Θα ψηφίσουμε επί των φακέλων όπως αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη. Η ψηφοφορία θα διαρκέσει από τις 9 ως τις 10 και 15. Θα χρησιμοποιηθεί η ίδια μέθοδος ψηφοφορίας που χρησιμοποιήθηκε και στις προηγούμενες ψηφοφορίες. Όλες οι ψηφοφορίες θα πραγματοποιηθούν με ονομαστική κλίση κηρύσω την έναρξη της πρώτης ψηφοφορίας. Μπορείτε να ψηφίσετε ως τις 10 και 15. Τα αποτελέσματα της πρώτης ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν στις 12 και 45. Σας ευχαριστώ.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 Επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση. Προχωρούμε στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της σημερινής πρώτης ψηφοφορίας. Έχουν ως εξής. Τελική ψηφοφορία για την έκθεση Ουρτάσουν ισότητα ανδρών γυναικών ε, στα πλαίσια εξωτερική πολιτική Ευρωπαϊκή Ένωση εγκρίθηκε ω είχε το σχέδιο ψηφίσματο. Ερχόμαστε στι τροπολογίε ε, τη έκθεση Αντριού για την κοινή γεωργική πολιτική. επί της ουσίας αρμόδια. Η Επιτροπή έχει τροπολογίες που εγκρίθηκαν κατά σύνολο. 10 εγκρίθηκε, 56 εγκρίθηκε, η 58 απερίφθη, τροπολογία 75 εγκρίθηκε, τροπολογία 76 εγκρίνεται, τροπολογία 102 το πρώτο μέρος εγκρίνεται, τροπολογία 102 δεύτερο μέρος εγκρίνεται, τροπολογία 120 πρώτο μέρος εγκρίνεται. Η τροπολογία 122 μέρος εγκρίνεται. Τροπολογία 132 απορρίπτεται. Τροπολογία 171 εγκρίνεται. Τροπολογία 205 πρώτο μέρος εγκρίνεται. Τροπολογία 205 δεύτερο μέρος εγκρίνεται. Τροπολογία 212 εγκρίνεται. Τροπολογία 266 εγκρίνεται. Τροπολογία 232 εγκρίνεται. Η τροπολογία 274 αναθεωρημένη απορρίπτεται. Η τροπολογία 257 εγκρίνεται. Τροπολογία 267 CP1 απορρίπτεται. Τροπολογία 258 D εγκρίνεται. Τροπολογία 267 CP2 απορρίπτεται. Τροπολογία 259 εγκρίνεται. Τροπολογία 260 αναθεωρημένη εγκρίνεται. τροπολογία 261 εγκρίνεται. Τροπολογία 233 εγκρίνεται. Τροπολογία 234 εγκρίνεται. Καταπίπτει 71. Τροπολογία 275 πρώτο μέρος απορρίπτεται. Το δεύτερο συνεπώς καταπίπτει. Τροπολογία 262 αναθεωρημένη απορρίπτεται. Τροπολογία 72 εγκρίνεται. Τροπολογία 255 απορρίπτεται. Η αναθεωρημένη τροπολογία 235 εγκρίνεται. Οπότε και καταπίπτει η τροπολογία 79. Τροπολογία 80 εγκρίνεται. Η τροπολογία 81 εγκρίνεται. Τροπολογία 268 απορρίπτεται. Τροπολογία 82 εγκρίνεται. Η τροπολογία 236 εγκρίνεται και καταπίπτει η τροπολογία 84. Αναθεωρημένη τροπολογία 263 εγκρίνεται. Οπότε και καταπίπτει η τροπολογία 89. Τροπολογία 237 εγκρίνεται και καταπίπτει η τροπολογία 90. Η τροπολογία 269 εγκρίνεται και καταπίπτει η τροπολογία 109 και το πρώτο και το δεύτερο μέρος Η τροπολογία 270 απορρίπτεται, η τροπολογία 110 εγκρίνεται, η τροπολογία 231 απορρίπτεται, η τροπολογία 238 εγκρίνεται και καταπίπτει 114. Η τροπολογία 239 εγκρίνεται και καταπίπτει η τροπολογία 117. Αναθεωρημένη τροπολογία 276. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 240 εγκρίνεται. Η 241 επίσης εγκρίνεται. Η τροπολογία 242 εγκρίνεται. Και καταπίπτουν οι τροπολογίες 271 και 122. Τροπολογία 272D απορρίπτεται, τροπολογία 123 εγκρίνεται, τροπολογία 243 εγκρίνεται, η τροπολογία 273 εγκρίνεται. Συγγνώμη, απορρίπτεται. Η τροπολογία 126 εγκρίνεται. Η τροπολογία 244 εγκρίνεται και καταπίπτει η τροπολογία 128. Τροπολογία 245 εγκρίνεται, οπότε και καταπίπτει η τροπολογία 129. Η τροπολογία 246 εγκρίνεται. Η αναθεωρημένη τροπολογία 277 απορρίπτεται. Η τροπολογία 150 εγκρίνεται. Τροπολογία 247 εγκρίνεται. Τροπολογία 248 εγκρίνεται. Τροπολογία 249 εγκρίνεται. Καταπίπτουν συνεπώς οι 153 και οι 154. Η τροπολογία 250 εγκρίνεται. Καταπίπτει 158. Η τροπολογία 264 απορρίπτεται, η τροπολογία 165 απορρίπτεται, η τροπολογία 254 απορρίπτεται, η τροπολογία 278 εγκρίνεται, η τροπολογία 251 εγκρίνεται, καταπίπτουν οι τροπολογίες 180 και 181. Η τροπολογία 252 εγκρίνεται, η καταπίπτει η τροπολογία 183 και 184. Τροπολογία 253 εγκρίνεται, καταπίπτει τροπολογία 187 όπως και 188. Τροπολογία 229 απορρίπτεται. Η τροπολογία 3 εγκρίνεται. Η τροπολογία 265 απορρίπτεται. Η τροπολογία 279 απορρίπτεται. Η τροπολογία 280 απορρίπτεται, η τροπολογία 230 απορρίπτεται, η τροπολογία 8 εγκρίνεται και τέλος η τροπολογία 256 εγκρίνεται. Διακόπτεται η συνεδρίαση μέχρι τις 1 και 4, οπότε και θα αρχίσει ο επόμενος γύρος ψηφοφορίας. an intervention in Der Präsident! Die Sitzung ist. Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται. Θα προχωρήσουμε στη σημερινή δεύτερη ψηφοφορία. Θα ψηφίσουμε από τον φακέλων όπω αναφέρονται στην μισή διάταξη. Η ψηφοφορία θα διαρκέσει από τη 1 και 4 έω τι 2.30 θα χρησιμοποιηθεί η ίδια μέθοδο ψηφοφορία που χρησιμοποιήθηκε και στι προηγούμενε ψηφοφορίε. Όλε οι ψηφοφορίε θα πραγματοποιηθούν με ονομαστική κλίση. Κυρίσω την έναρξη τη δεύτερη ψηφοφορία. Μπορείτε να ψηφίσετε έως τι 2.30. 14 και 30. Τα αποτελέσματα τη δεύτερη ψηφοφορία θα ανακοινωθούν στι 17 στι 5. Η συνεδρίαση διακόπτεται. Thank you. I thank you. I, yes, I you. Sitzung Επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση. Περνάμε στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του δεύτερου γύρου των ψηφοφοριών. Έκθεση Γιά για την κοινή γεωργική πολιτική για την χρηματοδότηση των στρατηγικών από το ΕΠΑ. Η πρόταση της ε, Κομισιόν, ε, όπως έχει τροποποιηθεί, γίνεται δεκτή. Όσον αφορά την έκθεση για υπάρχει το θέμα της αναπομπής, ε, η οποία επίσης γίνεται δεκτή. Μετά έχουμε έκθεση Μίλλερ για την κοινή γεωργική πολιτική, όσον αφορά την χρηματοδότηση και επιτήρηση των προτάσεων της Κομισιόν, όπως αυτές τροποποιήθηκαν, γίνεται δεκτή και έχουμε την έκθεση Μίλλερ επίσης ε, περί αναπομπής ε, και αυτό έγινε δεκτό. Και τέλος, έκθεση Αντριέ, κοινή γεωργική πολιτική για τον κοινό οργανισμό αγοράς και λοιπούς κανονισμούς ε, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν γίνεται δεκτή και η αναπομπή στην Επιτροπή επίσης. τα πρακτικά των ε, των συνεδριάσεων ε, της 19ης ε, και 20ης έχουν υποβληθεί για έγκριση και τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών θα διαβαστούν αρμοδίως. Τέλος, ζήτησα τον πρόεδρο να κάνω την εξή δήλωση. Θα ήθελα εξ ονόματός μου και των υπολείπων ε, συναδέλφων να ευχαριστήσω τους συναδέλφους, τους υπαλλήλους του Κοινοβουλίου που επιτρέπουν την διεξαγωγή της σημερινής συνεδρίασης ε, και των λοιπόν συνεδριάσεων. Χωρίς σας δεν θα είχαμε την δυνατότητα να ασκήσουμε πλήρως τα καθήκοντά μας, να νομοθετούμε και να υπηρετούμε τους πολίτες και να έχουμε στο επίκεντρο της δημοκρατίας. Σας ευχαριστώ για την δουλειά σας, τον επαγγελματισμό και την αφοσίωσή σας. Αυτά από εμένα και τον πρόεδρο. Η συνεδρίαση διακόπτεται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.